της πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Θα μας μιλήσει για την ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία. Έχετε το λόγο κυρία Μογκερίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζούμε σημαντικές στιγμές για την Πολωνία. Κολομβία. Ζούμε σημαντικές στιγμές για την, για την Κολομβία. Νομίζω ότι είναι μια περιοχή του κόσμου που έρχονται μηνύματα ελπίδας, μηνύματα αλλαγής και είναι καλό που οργανώνεται η συζήτηση αυτή γιατί είμαι πεπισμένη ότι αυτή τη χρονιά θα ακούσουμε νέα καλά, νέα ενδιαφέροντα μετά από πάρα πολλά χρόνια. 200.000 και άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από ένα εκατομμύριο εκτοπίστηκαν ουσιαστικά, μετακινήθηκαν χωρίς τη θέλησή τους, εκατομμύρια έπεσαν θύματα βίας, Οι διαπραγματεύσεις αυτές ε, ξεκίνησαν πάνω από ένα χρόνο και βλέπουμε ότι στην Αβάνα υπάρχουν κάποια μηνύματα θετικά. Είναι μηνύματα ειρήνης, είναι μηνύματα ελπίδας, είναι νέα καλά. Όπως ακούσαμε και στη Βιέννη για το Ιράν πριν μερικές μέρες. Είναι μια καλή ευκαιρία. Παρακολούθησα όπως φαντάζεστε ε, την ειρηνευτική διαδικασία ακόμα και πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις αυτές στην Αβάνα. Σαν υπουργό είχα επισκεφθεί την Πογκοτά και υποστήριξα τον τότε ε, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην τεράστια προσπάθεια την οποία έκανε. Νομίζω ότι τώρα υπήρξε ενίσχυση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ε, Κολομβία, υπήρξε η άδεια για την χορήγηση των θεωρήσεων, Προσπαθούμε να αποδείξουμε λοιπόν την προσπάθεια την συνεχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ειρηνευτικής διαδικασίας και οι τελευταίες αποφάσεις ελήφθησαν με πλήρη στήριξη και του Προέδρου Σάντος. Νομίζω λοιπόν ότι και οι εμπειρίες τις οποίες είχαμε από αντίστοιχες ειρηνευτικές διαδικασίες όπως αυτή της Ιρλανδίας ήταν ιδιαίτερως θετικές και είχαμε πάρα πολλές ε, μορφές ενίσχυσης των συναντήσεων. Ξέρω ότι ε, θα συναντηθεί ο πρόεδρος της χώρας ε, και με τα μέλη της Επιτροπής ΑΦΕΤ στο τέλος του μήνα θα παρουσιάσει τις δυσκολίες και τις ευκαιρίες της ειρηνευτικής διαδικασίας και θα συζητήσει με τα μέλη της Κοινοβουλευτικής σας Επιτροπής τις μορφές ενίσχυσης ε, της διαδικασίας. Λοιπόν, είμαστε, είμαστε στη βάση, εργαζόμαστε στη βάση της ε, συμφωνίας ε, για τα θύματα στην οποία είχαμε καταλήξει πριν μερικούς μήνες. Προήμιο για τη συμφιλίωση είναι η συμφιλίωση η μοναδική βάση θα έλεγα για να προχωρήσει η διαδικασία αυτή με αηφόρο τρόπο. Στην ουσία γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία γύρω από τη σύγκρουση αυτή, τις αιτίες, ε, τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί και την ανάγκη να μην επαναληφθούν. Επίσης πρέπει να γίνει προσπάθεια και για τους εξαφανιστέντες είναι σημαντικό για αυτούς οι οποίοι έχουν χάσει τους αγαπημένους τους να γνωρίζουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει και να τεθεί και το θέμα των αποζημιώσεων προς τα θύματα, είτε συλλογικά είτε ατομικά. Είναι πρώτη φορά που μια τέτοια συμφωνία παίζει κεντρικό ρόλο σε διαπραγματεύσεις ειρηνευτικές. Έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί υπάρχει από ό,τι φαίνεται μια νέα μορφή αντίληψης που θα επιτρέψει να γεφυρωθούν οι διαφορές. θα πρέπει από τη μία η ατιμορρησία να αποκλειστεί και ταυτόχρονα από την άλλη θα πρέπει να υπάρξει η ειρήνευση. Είναι μια ισορροπία δύσκολη αλλά οι Κολομβιανοί είναι πεπισμένοι ότι θα το πετύχουν. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι προτεραιότητα, ενίσχυση των δικαιωμάτων αυτών. Πολλές φορές αυτοί που τα προασπίζονται έχουν πέσει και συνεχίζουν να πέφτουν θύματα βίας και απειλών η Κολομβία έχει ξεκινήσει από μια πολύ δύσκολη κατάσταση, τα τελευταία χρόνια όμως έχει επιτελέσει σημαντικά βήματα προόδου, οι δυσκολίες υπάρχουν, αλλά και οι προσπάθειες που γίνονται θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση και ενίσχυση της ειρήνης. Δεν έχουν φυσικά ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις στη Σαββάνα. οι διαπραγματεύσεις αυτές συνεχίζονται, πολύ σημαντικά θέματα μένουν ακόμα προς διευκρίνηση όπως η συμφωνία, η εφαρμογή της, ο έλεγχος της, οι εγγυήσει για την ασφάλεια των φυσικών προσώπων που έχουν εμπλακεί στη σύγκρουση. Είμαι πεπισμένη πάντως ότι οι διαπραγματεύσεις θα ολοκληρωθούν και μάλιστα θα ολοκληρωθούν με αρκετά μεγάλη ταχύτητα σύμφωνα με τις ανηλυμένες υποχρεώσεις του Προέδρου Σάντους θα πρέπει να δούμε και ποια θα είναι η επόμενη φάση, πώς θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε εμείς την ειρήνη η οποία τώρα διαφαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει. Η εμπειρία δείχνει ότι η εφαρμογή μιας ειρηνευτικής δυσφωνίας είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Νομίζω ότι απαιτείται να κυριαρχήσει η νέα αντίληψη που θα αντικαταστήσει τις παλαιές προκαταλήψεις. Θα πρέπει και οι δύο πλευρές να μην προβούν σε ε, προκλήσεις και να εφαρμόσουν με σοβαρό τρόπο τις υποχρεώσεις που θα αναλάβουν. Αυτή είναι και η δική μας προσπάθεια και η δική μας εντολή να, να, ενισχύσουμε την φάση της εφαρμογής με όλα τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Εμείς αυτή τη στιγμή υπογραφεί μια τέτοια συμφωνία και επικυρωθεί θα ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τις προσπάθειές μας και για το θέμα του ελέγχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τη βοήθεια που πρέπει να δοθεί στη χώρα για να προχωρήσει σε βαθύτατες αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές θα οδηγήσουν στην βιώσιμη ειρήνη και όχι απλά σε στιγμιαία ειρήνη θα στηρίξουμε την Πολωνία όπως το κάναμε και την Κολομβία όπως το κάναμε και στο παρελθόν και νομίζω ότι έτσι θα βοηθήσουμε τα εμπλεκόμενα μέρη να πετύχουν τους στόχους τους. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και ένα καταπίστευμα το οποίο θα χρηματοδοτηθεί και από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και από τα κράτη-μέλη για την οικονομική ενίσχυση της χώρας. Προχωράμε στις προκαταρτικές εργασίες για την δημιουργία του καταπιστεύματος αυτού, για το οποίο υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα συμπληρώσει μια τέτοια προσπάθεια και τις προσπάθειες της ίδιας της ε, Κολομβίας σε οικονομικό επίπεδο. Εμείς δεν προσφέρουμε μόνο προθέσεις καλές, αλλά μια συνεχή πολιτική στήριξη την οποία οι Κολομβιανοί έχουν ανάγκη έτσι ώστε η ειρηνευτική αυτή διαδικασία όπως είπα να είναι βιώσιμη αυτή στιγμή υπογραφή και να συνεχιστεί τις επόμενες δεκαετίες. Θα συνεργαστούμε με τους διεθνείς εταίρους μας και στον τομέα της οικονομικής βοήθειας και θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε στην προσπάθεια επιτυχίας της Κολομβίας. Είναι σημαντικό το παράδειγμα αυτό γιατί η Αμερική είναι μια αλλαγή απαραίτητη που θα οδηγήσει στη συμφιλίωση. Αυτή η αλλαγή πρέπει να συνοδευτεί, να ενθαρρυνθεί και να ενισχυθεί. Πρόκειται για μια αλλαγή επιτέλους θετική και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάθε συμφέρον να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Όχι μόνο στην Κολομβία αλλά και στην Κολομβία γιατί όπως είπα εμείς προσπαθούμε να διαχειριστούμε τις κρίσεις γύρω από την Ευρώπη αλλά δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε τα θετικά βήματα τα οποία συμβαίνουν σε διάφορα σημεία του κόσμου που σταθεροποιούν την κατάσταση και οδηγούν σε πιθανές αλλαγές σε συγκρούσεις που κρατούν εδώ και δεκαετίες. Ακόμα και σε μακρινές αποστάσεις τέτοιες συγκρούσεις επηρεάζουν αρνητικά τον υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε κάθε λόγο λοιπόν να στηρίξουμε και να διευκολύνουμε με κάθε προσπάθεια την οποία πρέπει να κάνουμε την ειρηνευτική διαδικασία και σε πολιτικό και σε οικονομικό επίπεδο. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Αντιπρόεδρο. Ε, θα ακούσουμε λοιπόν τώρα την ε, άποψη των πολιτικών κομμάτων για αυτά που μας είπατε εκ μέρους του ΕΛΚ, ε, Γκράντε Πασκουάλ, για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε, είπατε εκπρόσωπε, κυρία Μογκερίνη. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω αυτά που εκτενώς περιέγραψε η κυρία Μογκερίνη σωστά και με ακρίβεια και με σοβαρότητα. Άξε τον κόπο γιατί είναι σήμερα ιστορική στιγμή. Εγώ θα μιλήσω τώρα με μια αξιολόγηση. Κατά την άποψή μας ε, το αξίζει η Κολομβία αυτό, αυτή την υποστήριξη. Με τη συμπεριφορά της το κατέκτησε. Και το λέω αυτό με κάθε επισημότητα. Είναι ιστορική στιγμή. Είχε όμως και προηγούμενα. Το προσπάθησαν και άλλοι. Υπήρξαν και άλλες απόπειρες με διάλογο μεταξύ ανταγωνιστικών ομάδων βρέθηκαν κάποιες λύσεις. Θυμίζω ότι πριν το Σάντος, η Μπερτανκούρο, Γκαβίρια, Όπαστα, ανά και ο ίδιος ο Ουρίμπε, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ο πρόεδρος Σάντος, εάν ολοκληρώσει αυτή την ιστορική ενευτική διαδικασία θα έχει ένα απόλυτο βάθρο που του αξίζει πραγματικά στην ιστορία της Κολομβίας να δούμε ποιε είναι οι συνθήκες Το Κοινοβούλιο που τόσο διαφέρει, που τόσο πολυφωνικό είναι, κατάφερε να περάσει ένα ψήφισμα επτά μεγάλων πολιτικών ομάδων με συνένεση και το οποίο μονοσήμαντα λέγει ότι κατά πλειοψηφία θα υποστηρίξει το ψήφισμα με τις αρχές και τις αξίες που πιστεύουμε ότι είναι στο ύψος των περιστάσεων. Πιστεύω ότι η Κολομβία το κέρδισε αυτό με τη συμπεριφορά τη Έκανε τη διαφορά. Τι λείπει τώρα κυρία Μογκερίνη. Αυτό που είπαμε και είπατε κι εσείς. Πόροι τώρα για να συνοδευτεί η νευτική διαδικασία η οποία αποκορυφώθηκε με μια δικαιοσύνη που δεν θα επιτρέψει ατιμορρησία, ε, θα υπάρξει ισότητα και θα επιτρέψει η Κολομβία να ζήσει αυτή την ιστορική τη στιγμή που χωρί καμιά αμφιβολία τη αξίζει και όλοι θα βοηθήσουμε να συναντήσει τη μοίρα τη. Ευχαριστώ. Να σέβεστε όλοι παρακαλώ τους χρόνους σας. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος ε, Χάουρεγγι Ατουόντο για δυόμιση λεπτά. Παρακαλώ Ραμόν, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Μογκερίνη πάρα πολύ για την παρουσία σας, για τα λόγια σας. Θα ήθελα να σας πω καταρχάς το εξή. Όπως γνωρίζουμε όλοι, η ανθρωπότητα ήδη εδώ και καιρό έχει καταδείξει ότι το τέλος ενός πολέμου είναι πολύ πιο δύσκολο από την αρχή του. Εσέδειξε η ανθρωπότητα ότι η διαπραγμάτευση με ε, μια τρομοκρατική οργάνωση για το τέλος της βίας είναι πολύ πιο δύσκολη από την αστυνομική ακόμα καταστολή και την πάταξη και τον πόλεμο προς μια τρομοκρατική οργάνωση. Όπως είπατε αυτά τα δύο μεγάλα επιτεύγματα και οι κατακτήσεις της Κολομβίας τους επόμενους μήνες πραγματικά σηματοδοτούν μια ιστορική στιγμή για την Κολομβία. Ας μην ότι μάλλον τώρα τερματίζουν αυτό που ήταν μια τραγική παράδοση για τη χώρα, πάνω από 50 ετών. Όχι μόνο στην Κολομβία, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες της Νοτιού Αμερικής, Κεντρικής Αμερικής, που επί σειρά ετών πολλές πολιτικές ομάδες θεώρησαν ότι η βία δικαιολογείται και νόμιμοποιείται για να φτάσουν στους πολιτικούς τους στόχους και σκοπούς. Σήμερα πιθανότατα είμαστε στο τέρμα αυτής της τραγικής ιστορίας και του τραγικού σφάλματος. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ποτέ δεν υπήρχαν λόγοι που να δικαιολογούσαν το να σκοτώνεις, το να ε, ε, χρησιμοποιείς τη βία. Πιστεύω ότι η απόφαση της Κολομβίας είναι αξιέπαινη έχει τεράστια σημασία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα μπορούσε να απέχει από αυτή. Όπως είπε και ο κύριος Δεγκράντες, ελάβαμε μια απόφαση σημαντική και επίκαιρη. Πάρα πολύ επίκαιρη, διότι μπορεί να έρθει η ειρήνη σε λίγους μήνες οριστικά. Και επίσης έχουμε δεσμευτεί, διότι συζητήσαμε για ε, τα όσα έχουν συμβεί στην Ευρώπη και δεσμεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διάφορες πολιτικές ομάδες να βοηθήσουν. Και είναι και γενναία αυτή η απόφαση διότι ομόφωνη και για πρώτη φορά σε ένα θέμα διεθνούς πολιτικής αποφασίζουμε ομόφωνα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέρ της συνευτική διαδικασίας. Μπορεί να μην είναι τέλεια η ειρήνη. Γνωρίζουμε ότι πολλοί είναι και αντίθετοι. Αλλά είναι ειρήνη. Γι' αυτό έχει σημασία να θυμίσουμε ότι δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος, όπως το έλεγε και ο Δάντης. Είναι πολύ σημαντικό να συναντήσουμε την ειρήνη που ε, λύθηκαν πολλά προβλήματα. Είναι σπουδαία είδηση και αξίζει την υποστήριξή μας και πολύ ωραία το είπε ε, ε, για το καταπίστευμα η κυρία Μογκερίνη και για ο διορισμός του κυρίου Γκίλμορ είναι πάρα πολύ σημαντικό. σημαντικός. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μογκερίνη. Ο κύριος Ντεμές Μάκερ για ένα λεπτό εξ ονόματος ε, των συντηρητικών. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, μπορούμε ακόμα να είμαστε αισιόδοξοι, στραμμένοι προς το μέλλον. Είναι διάφορες οι κρίσεις που σοβούν ανά την Ιφίλιο και μας κάνουν να αμφιβάλλουμε. Αλλά στην Κολομβία η πρόσφατη ενευτική διαδικασία με τους ΦΑΡΚ μας κάνει να ελπίζουμε ε, ότι κάποια στιγμή θα δούμε το τέλος του τούνελ. Μυρίζει άρωμα ειρήνης. Ε, τα, οι συμφωνίες, ε, οι προσωρινές θα ολοκληρωθούν στις 23 Μαρτίου και θα οδηγήσουν ε, στην παράδοση των όπλων του ΦΑΡΚ. Στο ψήφισμα της ομάδας μας εμείς καλούμε τα διάφορα μέρη στο μεταξύ να διασκεδάσουν όλες τις αμφιβολίες για τη μεταβατική δικαιοσύνη και να αποκατασταθούν τα θύματα. Η ενευτική διαδικασία όμως δεν μπορεί να σταματήσει εδώ. Υπάρχει και η βία του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού και των παραστρατιωτικών ομάδων ε, δεν συμμετείχαν οι παραστατιωτικοί όμως στη διαδικασία ένταξης μετά την αποστράτευση και φοβάμαι ότι οι παραστρατιωτικές ομάδες παραμένουν ε, και αντιμάχονται και την κυβέρνηση και ε, το στρατό δηλαδή της Ένωπης Δυνάμης αλλά και της ΦΑΡΚ. Θα πρέπει και αυτά να αντιμετωπιστούν. Ευχαριστώ κυρία Μπιλμπάο για 1,5 λεπτό. Ξέρω με τους Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα ξεκινώντας να συγχαρώ την προσπάθεια την οποία έχουν κάνει τα εμπλεκόμενα μέρη στην Κολομβία η απόδοση δικαιοσύνης και η αποζημίωση και αποκατάσταση των θυμάτων θα οδηγήσει στη μια επανάληψη αυτών των ενεργειών. Οι Κολομβιανοί και τα θεσμικά τους όργανα και η κοινωνία γνωρίζει πάρα πολύ καλά το κόστος του πολέμου και αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με πραγματισμό και θα πρέπει να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή. Θα πρέπει να δώσουμε παραδείγματα σε σχέση με το πώς μπορούμε να συνοδεύσουμε την προσπάθεια αυτή και εδώ αναφέρομαι και σε αυτά που είπε η κυρία Μόγκερίνη μέσω της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και τη συγχαίρω γι' αυτό. Έτσι θα μπορέσουμε να ε, μετατρέψουμε σε πραγματικότητα και τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες που έχουν γίνει και για την καταδίκη της βίας, για τη στήριξη της προσπάθειας πολιτικής λύσης, έτσι ώστε σε όλο τον κόσμο να μην υπάρχει α, στήριξη στην ατιμορρησία για εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας. Μια υποστήριξη λοιπόν στα θύματα, μια στήριξη στα θεσμικά όργανα, μια στήριξη στην κοινωνία, για σωστή πορεία, ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη και τελικά συμφιλίωση και όχι η διπλή θυματοποίηση της Κολομβίας αυτής. Η ταυτότητα της χώρας είχε ταυτιθεί με το αίμα, με την βία, με την κρίση και αυτό οδήγησε σε πάρα πολύ μεγάλη απώλεια αξιοπιστίας στο εξωτερικό. Η Κολομβία λοιπόν αλλάζει και περνάει από μια, σύγκρου, από μια χώρα με συγκρούσεις σε μια χώρα με ευκαιρίες. Κόζο περμούι από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ΚΟΕ ε, θα ήθελε και αυτή ε, να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να συνοδεύσουμε την διαδικασία αυτή την ειρηνευτική που θα θέσει τέλος σε 279.000 θύματα μέχρι τώρα, χιλιάδες συνδικαλιστές δολοφονημένους, πάρα πολλά θύματα από την κοινωνία των πολιτών, 6 εκατομμύρια ανθρώπων που έχουν ε, μετακινηθεί από τις αστείες τους με τη βία και νομίζω ότι οι προσπάθειες τις οποίες έχει κάνει και το ΦΑΡΚ και η Κολομβιανή κυβέρνηση και για τα θέματα της συμφωνίας για τα θύματα και για το θέμα που αφορά την εμπορία των ναρκωτικών είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να οδηγήσει και στην λαϊκή στήριξη της συμφωνίας αυτής με βάση την αλήθεια, με βάση τη δικαιοσύνη, με στόχο την προσπάθεια μη επανάληψης. Θα πρέπει επίσης να αφοπλισθούν οι πολιτοφυλακές οι οποίες είναι σε, εξυπηρετούν τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας, πολλές φορές και ευρωπαϊκών συμφερόντων, να προστατεύσει η Πολωνία επιτέλους τον πληθυσμό της, να προστατεύσει τα συνδικαλιστικά κινήματα, τα πολιτικά κινήματα, να υπάρξει λειτουργία και της υπηρεσίας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ και να στηρίξουμε και οικονομικά την χώρα αυτή μέσω των μηχανισμών διεθνούς αναγνώρισης. Ευχαριστώ κύριο Σεμπαστιά από πλευρά των Πρασίνων για 1,5 λεπτό. Σας... ευχαριστώ κύριε κυρία Μογκερίνη που ήρθατε εδώ για να πάρετε το λόγο αλλά και να μας ακούσετε. Είναι μια ευτυχή στιγμή. Θα πρέπει νομίζω να σας συγχαρούμε για τις προσπάθειες τις οποίες έχετε κάνει και για όλους όσους συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για τη συνεισφορά τους στην ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις τεράστιες προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων μερών θα πρέπει να εμπλακεί ακόμα περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση και στον εμπορικό τομέα, στις εμπορικές συμφωνίες. Θα πρέπει επίσης να δώσουμε και βοήθεια έτσι ώστε να βοηθήσουμε τον κόσμο που έχει αποφέρει. Θα πρέπει να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει επίσης να εμπλακούμε και στα πλαίσια της δημιουργίας ενός καταπιστεύματος από πλευράς των κρατών μελών για να βοηθηθούν τα θύματα της σύγκρουσης. Όπως είπε και ο προλαλής σας συνάδελφος, ε, οι εγκληματικές ενέργειες ε, των ε, παραστρατιωτικών ομάδων θα πρέπει να τερματιστούν και να διαλυθούν και να αφοπλιστούν οι ομάδες αυτές. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ναι μεν θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία συνολική αλλά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μην στηρίξουμε την ειρηνευτική διαδικασία. Ευχαριστώ κύριο Κοράο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα στην ε, υπατή εκπρόσωπο. Ε, συμφωνούμε λοιπόν με την υποστήριξη αυτού του ψηφίσματος ε, γιατί όπως ε, ακούσατε ήδη έχουμε να κάνουμε με μια ιστορική μοναδική στιγμή μια στιγμή από την οποία ξεκινάει μια νέα εποχή για την Κολομβία μια νέα εποχή όπου πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτό που με ανησυχεί εμένα είναι τι θα γίνει αύριο γιατί η διαδικασία της ε, ειρήνης είναι μια καλή συμφωνία αλλά όμως ε, δεν λαμβάνει υπόψη πολλά πράγματα όπως ε, παραδείγματο χάρη την αποζημίωση των θυμάτων πού θα βρεθούν τα χρήματα ή πάρα πολλά άλλα θέματα που έχουν παραμείνει ανεπίλητα. Αυτά δεν τα αναφέρουμε στο ψήφισμα διότι βεβαίως ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε να δώσουμε ένα θετικό μήνυμα. Εγώ όμως θεωρώ ότι αυτά θα δημιουργήσουν πρόβλημα στο μέλλον Γι' αυτό λοιπόν με μεγάλη χαρά δεχόμαστε αυτή τη νέα ιστορία, τη νέα τη ιστορία, αλλά γνωρίζουμε ότι πρέπει να δουλέψουμε σκληρά στο μέλλον για την Κολομβία. Μίλα Μουν, 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η Κολομβία ζει μια κρίσιμη φάση στην ιστορία της, όπως υπόθηκε πρόσφατα. Στην Αβάνα επαναλήφθηκαν οι ε, διαπραγματεύσεις για την οριστική συμφωνία πριν τις 20 Μαρτίου. Ποιος είναι ο στόχος? Να τερματιστούν ε, πάνω από 50 χρόνια σύγκρουσης και πολέμου που προκάλεσαν πολλά δεινά, πολλά θύματα θανάσου, θανάτους, ε, τεράστιες ε, εκτοπίσεις. Είναι πολύ σημαντικές οι σχέσεις μας με την Κολομβία και έχουν συσφιχθεί πρόσφατα τα τελευταία χρόνια. Η κυρία Μογκερίνη μίλησε για την πολυμερή εμπορική συμφωνία που ε, δείχνει θετικά αποτελέσματα. Έτσι ώστε για την Κολομβία η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο δεύτερος εμπορικός εταίρος παγκοσμίω. τονίζω το μεγάλο ρόλο που έχει παίξει και το Κοινοβούλιο για να καταφέρει αναφέρουμε την άρση θεωρήσεων διαβατηρίων για τους πολίτες της Κολομβίας. Τις 2 Δεκεμβρίου υπογράφηκε η συμφωνία και δείχνει πώς θέλει να δώσει όθηση στη σχέση της η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Κολομβία και με τους πολίτες της. Το Κοινοβούλιο μας αύριο θέλει να βοηθήσει στην αποκορύφωση τη συνευτική διαδικασία και τα κράτη-μέλη μαζί με την Ένωση να βοηθήσουν και στο καταπίστευμα που θα έρθει να συνοδεύσει την περίοδο μετά τη σύραξη. Βρισκόμαστε σε μια ιστορική, επαναλαμβάνω, ε, ε, περίοδο. Θέλει να βγει από την επικίνδυνη σύραγγα της βίας η Κολομβία και είναι μεγάλη χώρα και πολύ σημαντική της Νότιας Αμερικής. Ο πρόεδρος ε, Σάντος μίλησε για ιστορικούς κύκλους βίας που κλείνουν οριστικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για την εθνική σκηνή αλλά και για τη διεθνή. Ευχαριστώ κύριο Χάου. Είτε 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, εγώ είχα την ευκαιρία να είμαι παρόν στην Αβάνα και να βοηθήσω και εγώ με την εμπειρία της δικής μου της χώρας σχετικά με την ειρήνευση στη Βόρεια Ιρλανδία. Ε, έχω λοιπόν σε όλη μου αυτή την κοινοβουλευτική θητεία αγωνιστεί για την Κολομβία και πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει ένα ιστορικό, μια ιστορική τομή. Ε, πριν από λίγο μια κοπέλα ε, δολοφονήθηκε και άλλοι ακτιβιστές ε, Βεβαίω η κυβέρνηση ε, κατόρθωσε να ε, αναστείλει απεργίες όμως απαιτούνται και πολλά άλλα πράγματα. Η συμφωνία ε, για τα θύματα είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα των κομμάτων και αυτό με έπεισε ότι τώρα πλέον ο δρόμος της ειρήνευσης ε, είναι χωρίς επιστροφή. Πρέπει και οι δύο πλευρές ε, να αναλάβουν την ευθύνη τους για την ειρήνη. Όσοι λοιπόν επιτίθενται στην ειρηνευτική διαδικασία για την περίφημη ατιμορρησία θα πρέπει να γνωρίζουν ότι παραμένει το ε, Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και αυτό νομίζω ότι θα μπορεί να δώσει κάποια ε, λύση στο πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει την ειρήνη και όπως έχει καταστήσει σαφές θέλουμε να ακολουθηθεί το μοντέλο της ε, Ιρλανδίας ή διαπραγματεύσει για την ειρήνη να είναι ανεξάρτητες με συμμετοχή και των δύο πλευρών και της κοινωνία των πολιτών. Επίσης να υπάρχουν και χέγγια ασφάλειας, η δημοκρατική αντιπολίτευση να είναι ανεξάρτητη, να μην επαναληφθεί η ε, σφαγή και σφαγές που έχουν λάβει η χώρα στο μέλλον να υπάρχει ειρήνη με δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη για την Κολομβία έχει φτάσει η στιγμή της ειρήνης. Ευχαριστούμε πολύ. κύριος Στυρ για 1,5 λεπτό. Παρακαλώ, έχει το λόγο κύριε Στυρ μετά από 50 χρόνια ένοπλης σύρεξη που έχει ξεκληρίσει ε, την Κολομβία και κόστισε πάνω από 200.000 ζωές έχουν αρχίσει τώρα μια συμφωνία για να δημιουργηθεί ειδική δικαιοδοσία για την ειρήνη που θα ε, δίνει ε, δικαίωση στα θύματα σε μια μόνιμη βάση και διαρκή. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συμφωνία, μπορεί να γίνει ιστορική εάν ολοκληρωθεί με επιτυχία. Γι' αυτό θέλουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφράσουμε την ικανοποίησή μα για τη συμφωνία του περασμένου Σεπτεμβρίου, αλλά θέλουμε να υποστηρίξουμε για να ε, κλείσει η οριστική συμφωνία πριν τι 23 Μαρτίου, που την έννοια αυτή η κυρία Μογκερίνη εσείς διορίσατε τον πρώην Ιρλανδό Υπουργό Εξωτερικών Σίμον Γκίλμορ, ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ευτική διαδικασία στην Κολομβία και σίγουρα αυτή η απόφαση ήταν πάρα πολύ εύστοχη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα θα πρέπει να εμβαθύνει την υποστήριξή της με ένα καταπιστευματικό ταμείο για την Κολομβία όπως προτείνουμε στο σχέδιο ψηφίσματος και χαιρόμαστε που εσείς μαζί με τον Επίτροπο Μίμητσα εργάζεστε προς την κατεύθυνση αυτή. Και είμαι Κροάτη εγώ όπω και ο επίτροπο Μίμητσα και γνωρίζουμε πολύ πόσο μεγάλη είναι η σημασία τη υποστήριξη τη διεθνού κοινότητας στι ε, διαδικασίε Θέλω να τονίσω και πάλι ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνοδεύει με τρόπο ενεργό σε αυτό το δρόμο την Κολομβία. Ευχαριστώ πολύ. Τζουρίνιο, δύο λεπτά. Πρόεδρε, κυρία Μογκερίνη, θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ για την προσπάθεια την οποία έχετε κάνει. Γνωρίζουμε ότι μια ειρηνευτική διαδικασία όπως αυτή της Κολομβίας είναι μια δύσκολη διαδικασία, είναι μια εύθραυστη διαδικασία και έχουμε καθήκον εμείς να προσπαθήσουμε όλες τις πλευρές να τις διευκολύνουμε. Θα πρέπει ταυτόχρονα αυτή η ειρηνευτική διαδικασία να συγκεντρώσει την προσοχή της όπως και προσπαθεί να το κάνει ε, στα θύματα και στις ανάγκες των θυμάτων. Συνεπώς λοιπόν η ειρηνευτική διαδικασία πρέπει να βοηθήσει όπως και έχει βοηθήσει μέχρι τώρα στην ε, ε, προσπάθεια αυτή. Η προσπάθεια που έχει γίνει όμως δεν είναι επαρκής γιατί πέραν της οικονομικής διάστασης η οποία θα πρέπει να οδηγήσει στην ενίσχυση της Κολομβίας θα πρέπει να αναλάβουμε και υποχρεώσεις για την εμβάθυνση της δημοκρατίας, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προσπάθεια να ζήσουν οι λαοί με ευμάρεια. Συνεπώς λοιπόν πρέπει να ενισχύσουμε μια ειρήνη βιώσιμη, πρέπει να ενισχύσουμε την κοινωνία των πολιτών, την ταλαιπωρημένη στην, στην Κολομβία, οι σχέσεις ανάμεσα στην Κολομβία και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει άλλωστε να αποτελέσουν και την σωστή πλατφόρμα για τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Νομίζω ότι το ψήφισμα του Κοινοβουλίου χαιρετίζει και την βούληση για συμβιβασμό και συνένεση όλων των εμπλεκομένων πλευρών. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την κουλτούρα της μη βίας στο εσωτερικό της κολομβιανής κοινωνίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δύναται και οφείλει να υποστηρίξει την ειρηνευτική διαδικασία ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ τον κύριο Τσουρίνιο. Υπάρχει μια μπλε κάρτα για σας από τον κύριο Άρνοτ. Δέχεστε την μπλε κάρτα. Ο κύριος Άρνοτ έχει το λόγο. Ζούμε σε ένα κόσμο όπου ε, συνεχώς ενημερώματα για τραγικές συγκρούσεις. Τα βλέπουμε αυτά σε καθημερινή βάση. Συμφωνείτε μαζί μου ότι η αχτίδα ελπίδας για χώρες όπως η Κολομβία ε, πολλές φορές ε, δεν καταγράφονται στα μέσα ενημέρωσης. Ίστες θα πρέπει να μην ξεχνάμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί καθώς προχωράει και ο κόσμος. Κύριε Τζουρίνιο, παρακαλώ την απάντησή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση. Κοιτάξτε, ε, πράγματι ε, κάθε μέρα ερχόμαστε αντιμετωπιμένες σε συγκρούσεις ε, και κάθε φορά που έχουμε να κάνουμε με ένα νέο πρόβλημα Αναφέρεται το πρόβλημα αυτό στα μέσα αλλά δεν αναφέρεται ποτέ η πρόοδο και από αυτού δεν μπορεί να ε, βρεθεί καμία λύση. Στην Κολομβία έχουμε, είχαμε μέχρι πρόσφατα πάρα πολλούς ε, θανάτους, νεκρούς, ε, αγνοούμενος. Ε, τώρα λοιπόν μετά την ε, διαδικασία που ξεκίνησε στην Αβάνα ε, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι πράγματι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα και αυτό που είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι ότι επιτεύχθηκε συμφωνία σε πολλά σημαντικά θέματα όπως στην αναδιάρθρωση της γης, σαν παράδειγμα το λέω, αλλά και σε πάρα πολλά άλλα. Μετά από όλο αυτό το κύμα βίας είναι σωστό να επισημάνουμε το ότι πρέπει να ληφθεί μέρημνα για τα θύματα. Το θέμα που τίθεται είναι πώς μπορεί κανείς να θεραπεύσει τις ε, πληγές. Ε, γιατί προβλέπεται ε, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα δικαιοσύνης. Ε, πρώτα απ' όλα όμως, ε, μέχρι τέλη Μαρτίου, θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια συνολική συμφωνία για να υπάρξει ε, εκεχηρία διαρκείας. Η Κολομβία είναι ένας από τους τελευταίους προμαχώνες των ιδεολογιών του προηγούμενου αιώνα και θέλω να σας πω ότι βλέπουμε ότι υπάρχει η επιρροή από όλους αυτούς που λένε ότι ε, δεν έχουμε την, ε, το δικαίωμα να επιτρέψουμε άλλο ένα πόλεμο, ας κάνουμε ό,τι μπορούμε να το επιτύχουμε. Ενάμιση λεπτό Δίας Δεμέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ ειλικρινά τον πρόεδρο Σάντος. Ο πρόεδρος Σάντος έδειξε γενναιότητα και ε, πήρε και κινδύνους. Ε, και κατάφερε με την τόλμη και τη γενναιότητα να φτάσει στη συμφωνία του Σεπτεμβρίου. Θέλω εδώ να τονίσω, όπως και άλλοι συναδελφοί, τη δημιουργία μιας ειδική προσωρινής δικαιοδοσίας για την ειρήνη, πολιτικής ε, γεωργικής ανάπτυξη ολοκληρωμένη, πολιτική, πολιτικής συμμετοχής και κάποια απάντηση στο ε, πρόβλημα των εκτοπισμένων, ε, ε, όλα αυτά ε, και τα θύματα και εκτοπισμένοι και οι γέες και τα άλλα ζητήματα χρειάζονται μεγαλύτερη προσήλωση. Ελπίζω στις 20 Μαρτίου να έχουμε οριστική συμφωνία και ελπίζω η Κολομβία να έχει την εμπιστοσύνη που της χρειάζεται και εσωτερική και εξωτερική και την αυτοπεποίθηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει στην Κολομβία και την εμπιστεύεται. Επανελειμμένα το έχει αποδείξει ο κύριος Γκίλμορ, ειδικό απεσταλμένος ε, για την διαδικασία. Εμπορική συμφωνία ή ακόμα και απελευθέρωση ε, θεωρήσεων. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα και παραδείγματα που δείχνουν ε, πόσο εκτιμούμε και βοηθούμε την Κολομβία. Έχει όμω ακόμα μεγάλη πρόκληση μπροστά τη υπενηχθήκατε την φάση μετά τη σύραξη και την οικοδόμηση της ειρήνης. Έχει σημασία εδώ η βοήθεια που μπορεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ε, έχει επίσης σημασία ε, το καταπίστευμα που θα συνοδεύσει αυτή την προσπάθεια να ευδοκιμήσει και πολλά ακόμα και μεταξύ αυτών η έναρξη διαπραγματεύσεων ε, με το Εθνικό Απελευθερωτικό Στρατό και άλλες παραστρατιωτικές δυνάμεις και πολιτοφυλακές που ακόμα διαταράσσουν την ειρηνική συνύπαρξη των Κολομβιανών. Ο κύριος Πέτερλε. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε το αποτέλεσμα της ε, ειρηνευτικής ε, διαδικασίας ε, είναι σημαντικό. Μόνο η ειρηνευτική διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε κάποια οριστική λύση του προβλήματος. Πλέον στην Κολομβία υπάρχει μια νέα πραγματικότητα και αυτή η πραγματικότητα θα απελευθερώσει ένα μεγάλο δυναμικό. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ τους πολιτικούς ηγέτες Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον Παπαφραγκίσκο και σε άλλους εμπλεκόμενους γιατί όλοι συνέβαλαν στο να υπάρξει ε, μία πολιτική λύση. Πρέπει να ανοίξει μία νέα σελίδα ε, στην Κολομβία προς όφελος ε, του λαού. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ η συμφωνία να υπάρξει ειδικό δικαστήριο για τα θύματα του πολέμου της Κολομβίας αυτή είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ειρήνης. Είχαμε χιλιάδες θανάτους, ε, ανθρώπους που πέθαναν από τα βασανιστήρια, από καταναγκαστικά έργα. Αυτά ήταν καθημερινότητα σε αυτή τη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν χαιρετίζουμε τη συμφωνία της Σαμπάνας του Δεκεμβρίου στο να υπάρξει ένα ειδικό δικαστήριο ε, που θα επιβάλλει την ειρήνη. Ελπίζουμε το 2016 να έχουμε την τελική και συνολική συμφωνία. Μετά την ε, πάψη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 Η Κολομβία είναι ένα πολύ δυσάρεστο παράδειγμα μιας κατάστασης όπου ορισμένοι πιστεύουν ότι μπορούν να επιβάλλουν με τη βία τους δικούς τους τους όρους. Όλα αυτά τα χρόνια τη ένοπλης σύγκρουσης δολοφονήθηκαν χιλιάδες άνθρωποι. Είχαμε 7 εκατομμύρια θύματα και αυτό είναι ανησυχητικό για πάρα πολλές χώρες του κόσμου αλλά και για πολλά πολιτικά κόμματα ακόμα και στην Ευρώπη. Ε, ανησυχητικά όλα αυτά για όσους ε, πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν την πραγματικότητα με τη βία ότι μπορεί κανείς ε, να ασκεί βία έναντι του ίδιου του, του κράτους. Οφείλουμε τέτοιου είδους παραδείγματα να τα αναφέρουμε ως κακά παραδείγματα και ε, χώρες όπως η Κούβα ας μην ξεχνάμε πρέπει να τις ευχαριστήσουμε ε, γιατί συνέβαλαν στο να επιτευχθεί η ειρήνη και ελπίζω επιτέλους να φτάσουμε σε μια οριστική ειρήνη. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα ξεκινά η διαδικασία Catch the Eye. Κύριος ε, Φαρία, παρακαλώ για ένα λεπτό. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το 2016 μπορεί να είναι μια πολύ αποφασιστική χρονιά για την Κολομβία με την πιθανή υπογραφή της ειρηνευτικής διαδικασίας που θα θέσει τέρμα σε μια σύγκρουση με τόσες χιλιάδες θύματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέκαθεν υποστήριζε τις ειρηνευτικές διαδικασίες και εξακολουθεί να υποστηρίζει σήμερα την κυβέρνηση του Πρόεδρου Σάντους θα πρέπει να υπάρξουν συνοδευτικά μέτρα τα οποία θα στηρίξουν την διαδικασία που έχει ξεκινήσει, θα πρέπει να ενισχυθεί η οικονομία της χώρας, θα πρέπει να μετατραπούν οι Γουεριέρος σε ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να περάσουμε λοιπόν από τη διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης για να οδηγηθούμε σε μια ειρήνη βιώσιμη. Ελπίζω, Πρόεδρε, ότι το Κοινοβούλιο μας θα βοηθήσει όσο μπορεί περισσότερο την Κολομβία να εμπλακεί στην οδό της δημοκρατίας αντίθετα με αυτά που συμβαίνουν στην Βενεζουέλα. Κύριος Χουαρίστη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Την ομάδα, η ομάδα μου ούτε εγώ δεν θα γράφω με αυτό το κείμενο αλλά χαίρομαι που το Κοινοβούλιο συζητά κοινή πρόταση για την ευτική διαδικασία στην Κολομβία και την υποστηρίζει. Θα πρέπει να χαιρόμαστε για όλα αυτά που πέτυχε η κυβέρνηση και η ΦΑΡΚ ήδη παρά τις δυσκολίες και τα απρόπτα και θα πρέπει επίση να συγχαρούμε και την κοινωνία τη Κολομβίας και να εθαρρύνουμε την κυβέρνηση και ε, το ΑΕΛΕΝ να ε, συνεχίσουν το διάλογο και να τον ολοκληρώσουν. Κυρία Μογκερίνη, κατά την άποψή μου, η ευρωπαϊκή βοήθεια δεν θα πρέπει να φτάνει μόνο στο κράτος της Κολομβίας, αλλά και στις επαρχίες και στις περιφέρειες, για να είναι εγγυημένη και η περιφερειακή ειρήνη. Θα ήθελα τέλος να τονίσω ότι είναι τουλάχιστον απορία άξιο που το Ισπανικό κράτο υποστηρίζει την ευτική διαδικασία στην Κολομβία και χαίρομαι γι' αυτό αρνείται να λυθεί δημοκρατικά η πολιτική σύγκρουση στη χώρα των Βάσκων. Θέλω να παροτρύνω όλους και όλες να εμπλακείτε και στη δική μου χώρα. Ευχαριστώ. Ε, έχετε μπλε κάρτα. Κύριε Χωρίστη. Από τον κύριο Ντεγκράντη Πασκουάλ. Τη δέχεστε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Χουαρίστη, πώς έχετε την ανέβεια να συγκρίνετε ένα διάλογο σε ένα δημοκρατικό κράτος που αναγνωρίζει τα λάθη του και κάποιες δυνάμεις που κάνουν ό,τι μπορούν. Και δεν θέλω να μπω στην ουσία. Ένα υποτιθέμενο διάλογο από μια τρομοκρατική δράση της ΕΤΑ με ένα ε, δημοκρατικό κράτος. Τέτοια ανέβεια, τέτοιο θράσος. Πού το βρήκατε. Ευχαριστώ κύριε Ντεγκράντης για την ερώτησή σας. Αυτό είναι κοινή λογική. Πολιτική σύγκρουση για οποιαδήποτε επίλυση πολιτικής διαφοράς έτσι γίνεται. Ο, ε, με, με, τη συζήτηση αυτό κάνετε και στην Κολοβία και χαίρομαι πάρα πολύ. Στην Ευρώπη, στην Ιρλανδία όπως το Κοινοβούλιο υποστήριξε την ευτική διαδικασία. Επίσης υπάρχουν και άλλες διαδικασίες που χρειάζονται την ε, θεσμική υποστήριξη της κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης τη συμμετοχή της δικής σας κυβέρνησης. Έτσι λύνονται οι πολιτικές συγκρούσεις. Είναι απολύτως απαραίτητο αυτό. Κύριε κύριος ένα λεπτό και εσείς παρακαλώ. Καλώς. Καταρχάς πιστεύω ότι ήταν σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στείλει ένα σημαντικό και κατηγορηματικό μήνυμα για την υποστήριξη της ενευτικής διαδικασίας. Αύριο θα γίνει και είναι πολύ θετικό βήμα. Θέλω να ευχαριστήσω και την ύπατη εκπρόσωπο για τα λόγια της και για τις προσπάθειες που κάνει για να συνοδεύσει αυτή τη διαδικασία. Πολύ σημαντικό. Το μόνο μήνυμα που θέλω εγώ να στείλω ε, είναι ότι δεν θα πρέπει να ε, εφησυχάσουμε ότι όλα γίνανε. Θα πρέπει οι συμφωνίε να υλοποιηθούν, αλλά απομένουν πολλά. Εμεί έχουμε πρόβλημα με του εκτοπισμένου, με τους ε, αυτόχθονες, με τι γυναίκε, με τι γέε. Έχουμε ε, γυναικοκτονίε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Κολομβία και δεν τα εξετάζουμε. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό, τα παραστρατιωτικά και οι πολιτοφυλακέ που πρέπει να διαλυθούν, να παραδώσουν τα όπλα. Είναι πολύ σημαντικό, Αλλιώ δεν υπάρχει ειρήνη που να στέκει. Και ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι η προστασία προστασία των ε, αγωνιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν υποφέρει τα πάνδυνα τα τελευταία χρόνια, υφίστανται τεράστιε διώξει και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το ξέρει αυτό. Σα παροτρύνω η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρακολουθεί και την ε, ολοκλήρωση και την κορύφωση και την υλοποίηση τη ε, ναυτική αυτή συμφωνία. Ευχαριστώ. Presidente. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στην Κολομβία επιτόλους ε, το σκοτάδι της σύραγγας είναι λιγότερο ε, πυκνό. Υπάρχουν λάθη στην ιστορία. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να λυθεί μια σύγκρουση που διαρκεί πάρα πολλά χρόνια. Έχουν αντιμετωπιστεί πολλά θέματα. Παραδείγματο χάρη όσον αφορά την ε, τον περιορισμό της ελευθερίας ε, θρησκευτικών απόψεων. Βεβαίως ε, ακόμα κρεμούν θέματα όπως το να αποσμιωθούν τα θύματα και πάρα πολλά άλλα συναφή. Και η συμμετοχή στην πολιτική ζωή για να μην μιλήσουμε για τις ε, τιμωρίες που πρέπει να επιβληθούν στους εμπλεκόμενους στον πόλεμο. Είναι σημαντικό να μην δοθεί αμνηστία στα σοβαρά εγκλήματα ε, να αντιμετωπιστεί το λατρεμπόριο των ναρκωτικών ε, γιατί τα θύματα είναι πραγματικοί πολίτες και δεν είναι συνομότες. Εξάλλου, εκ μέρου του Κολομβιανού κράτους ε, θα πρέπει να επιδιωχθεί σεβασμός των δικαιωμάτων όλων των πολιτών. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει και εμείς να σταθούμε στο ύψο μας των οικονομικών υποχρεώσεων, να δώσουμε στους νέους Κολομβιανούς την ελευθερία και να μην μάθουν ποτέ τι σημαίνει η λέξη πόλεμος. Κύριος για ένα λεπτό. Το τελικό στάδιο της ειρηνευτικής διαδικασίας ανάμεσα στην κυβέρνηση της Κολομβίας και τους αντάρτες του ΦΑΡΚ θα ολοκληρωθεί το Μάιο του 2016. Στις 15 Δεκεμβρίου υπογράφηκε συμφωνία για την αποζημίωση των θυμάτων του πεντηκονταετού πολέμου ανάμεσά του, ενώ οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για να μειωθούν οι επιχειρήσει του στρατού δρομολογούνται από το 2012 αρχικά με την ερευτική διαδικασία αναμένεται να σταματήσει η παλαιότερη και μεγαλύτερη σε διάρκεια διαμάχη στη λατινική αμερική που έχει τουλάχιστον 220.000 θύματα και έχει οδηγήσει σε πολιτικές διώξει τη αντιπολίτευσης και των συνδικαλιστικών ηγετών. παράλληλα προβλέπεται η αποζημίωση των θυμάτων τη διαμάχης καθώ και μέτρα για την καταπολέμηση τη διακίνηση των ναρκωτικών αλλά και για την ανάπτυξη τη αγροτική οικονομία. Επομένω, είναι αναγκαίο να ολοκληρωθούν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσει στην κολομβία ώστε να ξεκινήσουν έρευνε για του εξαφανιστέντε από την πολύχρονη διαμάχη καθώ και για να δημιουργηθεί ειδική επιτροπή που θα αποσαφηνίσει τα όσα συνέβησαν στον εμφύλιο πόλεμο. η ειρηνευτική διαδικασία άλλωστε μπορεί να οδηγήσει στη διαμόρφωση δημοκρατική κολομβίας υπό τον όρο ότι θα διαλυθούν οι παραστρατιωτικέ οργανώσει. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά κυρία Μογκερίνη. Σεβόμεθα ιδιαίτερα στην προσπάθεια που κάνουμε. Οι χιλιάδες θυμάτων και πάντα υπήρχε μια στρατηγική απόκρυψη της αλήθειας και υπήρχε επίσης και θεσμική βία όπως έχει αποδείξει η μελέτη του παρελθόντος. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο θα γίνει και σε σχέση με την μνήμη και σε σχέση με τον σεβασμό των θυμάτων απαιτείται δικαιοσύνη απαιτείται η ισότητα στην αντιμετώπιση και απαιτείται επίσης και απόδοση των ευθυνών. Νομίζω ότι στο προσεκτικό μας ψήφισμα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συμμετέχει στις διαδικασίες αυτές και το ποσοστό των θυμάτων που ανήκουν στην κοινωνία των πολιτών είναι άνω του 20%. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει να επικρατήσει η δικαιοσύνη και για την Κολομβία αλλά και για οποιοδήποτε μέρος στον κόσμο που παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ τερματίζεται η συζήτηση. Θα δώσω την ευκαιρία στην κυρία Μογκερίνη να δώσει την τελική καταληκτική της απάντηση. Να ξεκινήσω λέγοντας αυτό που είπατε ότι δεν έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία ακόμα αλλά είναι ένα μεγάλο μήνυμα ένα μεγάλο βήμα μάλλον έχουμε ξεπεράσει κάποιες πολύ δύσκολες στιγμές στις διαπραγματεύσεις αυτές νομίζω όμως ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτό ήταν επικοδομητικός και γι' αυτό υπογραμμίζω όπως είπα και στην εισαγωγή μου, ότι η υποστήριξή μας δεν αφορά μόνο την συνέχεια και την εφαρμογή της συμφωνίας, αλλά και τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες προσπαθούμε να συνοδεύσουμε τις διαπραγματεύσεις αυτές, να τις υποστηρίξουμε, να υποστηρίξουμε επίσης και την ηγετική προσπάθεια την οποία κάνει ο πρόεδρος Σάντος, ο οποίος έχει εντυπωσιάσει προς την κατεύθυνση αυτή, και να υποστηρίξουμε και το σύνολο της χώρας. Εγώ συμφωνώ σε αυτό το οποίο είπατε ότι θα πρέπει η υποστήριξή μας να φτάσει σε όλες τις περιφέρειες και σχετικά τώρα με ε, με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ είναι ένας ρόλος τον οποίο μπορεί να παίξουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα οποία έχουμε κάνει για την απελευθέρωση των θεωρήσεων ήταν πάρα πολύ σημαντικά γιατί όχι μόνο δείχνει τη στήριξη στην διαδικασία από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δείχνουμε ότι η προσπάθεια αυτή είναι ένα κομμάτι μιας ευρύτερης εικόνας του συνόλου των σχέσεων τις οποίες έχουμε με την Κολομβία και φυσικά αυτό εντάσσεται ακόμα περισσότερο και στο σύνολο των στρατηγικών σχέσεων που έχουμε με τη Λατινική Αμερική και τις οποίες αναπτύσσουμε με πολύ θετικό τρόπο ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Εμείς συναντηθήκαμε τις τελευταίες, ε, τους τελευταίους μήνες, τελευταία χρόνια, τεσσέρις-πέντε φορές ε, με ε, τον πρόεδρο Σάντος και με αφορμή την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Έχουμε τακτικές συναντήσεις, όποτε συναντώμεθα σε διάφορα φόρα στον κόσμο, πάντα συζητάμε είτε στην κορυφή για την Λατινική Αμερική, για, τη, τις δύο πλευρές μάλλον της Αμερικής. Προσπαθούμε, εν πάση περιπτώσει, να στηρίξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προσπάθειες ε, του Προέδρου και τις προσπάθειες της Κολομβίας. Νομίζω ότι έχουμε κάποια θετικά μηνύματα, έχουμε θετικές εμπειρίες και σε σχέση με τις εμπειρίες που έχει ο κύριος Γκίλμορ, ο διαπραγματευτής ε, από την Ιρλανδία και νομίζω ότι ε, οι δυσκολίες υπάρχουν αλλά προσπαθούμε να τις ξεπεράσουμε. Κάποιοι αναφερθήκατε στο παράδειγμα του τι μπορεί να κάνει και ποια μπορεί να είναι η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχάς αυτό είναι ένα δείγμα τις προσπάθειες την οποία κάνουμε ακόμα και σε περιφέρειες μακράν της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Είναι θέματα τα οποία αφορούν και τη δική μας όμως περιοχή, την δική μας περιφέρεια και τον Βορρά και τον Νότο θα πρέπει ακόμα και σε θέματα που έχουν σχέση με την Αρκτική ας πούμε και αυτό ακούγεται λίγο περίεργο από μια Ιταλίδα να το λέει, αλλά έχει σημασία να κάνουμε αυτό το οποίο μας αναλογεί και η προστιθέμενη αξία την οποία μπορούμε να προσδώσουμε είναι υψηλή ακόμα και στην Αφρική, ακόμα και στη Λατινική Αμερική, όχι παντού και πάντα, αλλά σε συγκεκριμένες περιοχές όπου η ιστορία, η πολιτική, η οικονομία, ο πολιτισμός βοηθά και υπάρχουν σύνδεσμοι, υπάρχουν σχέσεις που καθιστούν τις θέσεις μας χρήσιμες και πολύτιμες για τους πολίτες αυτών των χωρών. Αυτό είναι ο σφαιρικός ρόλος της Ένωσης, αυτή είναι η προσπάθεια την οποία θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ειρήνη στον κόσμο. Όταν το λέμε αυτό ακούγεται και ε, ίσως λίγο κενό αλλά παρόλα αυτά είναι προς όφελος όλων. Αυτός λοιπόν είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να επενδύσουμε σε αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να βγουν από τις συγκρούσεις. Είναι πιο δύσκολο να τερματίσει κανείς μια σύραξη παρά να ξεκινήσει μια σύραξη. Υπάρχει λοιπόν ένας τρόπος, ένας ευρωπαϊκός τρόπος για τη διευκόλυνση του διαλόγου, της συνεργασίας, της διαιτησίας, της διαμεσολάβησης και της συνένεσης. Αυτό ισχύει και για τις επόμενες συζητήσεις που θα κάνουμε, είτε ειδικά για τη Συρία, είτε συνολικά για τη Μέση Ανατολή. Η ευρωπαϊκή ιστορία με τους αιώνες συγκρούσεων μας έχει διδάξει πολλά έχουμε συμπαρασύρει πολλές φορές άλλους στους δικές μας συγκρούσεις, αλλά προσπαθήσαμε και θέσαμε τέλος σε αυτά μέσω ακριβώς της περιφερειακής συνεργασίας στην Ευρώπη. Και αυτό μας οδήγησε στην ειρήνη, την σταθερότητα και την ευημερία. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος, ο ευρωπαϊκός δρόμος Έχουμε μια καλή εικόνα στον υπόλοιπο κόσμο και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει τα καλά νέα από όπου και όταν ακούγονται. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τις ειρηνευτικές διαδικασίες όπου και αν συμβαίνουν. Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερο την ενότητα την οποία επιδείξατε κατά τη διάρκεια της συζήτησης και την οποία θα επιδείξετε είμαι βεβαία και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Και οι Κολομβιανοί φίλοι θα το κατανοήσουν, θα το αξιολογήσουν και θα το εκτιμήσουν. Και αυτό επίσης βοηθά μια δύσκολη διαδικασία αλλά δείχνει και την πολιτική μας υποστήριξη η οποία είναι πολύτιμη σε αυτές τις κρίσιμες μέρες. Ο Πάπας Φραγκίσκος είπε ότι η νύχτα της βίας μπορεί να γίνει μέρα αλλά η μέρα αυτή δεν θα πρέπει να έχει α, γρήγορη δύση. Θα πρέπει να βοηθήσουμε το δρόμο για την ειρήνη και τη συμφιλίωση. Αυτά τα λόγια του Πάπα Φραγκίσκου θα μας εμπνέουν. Θα συνεχίσουμε τις επαφές με τους κολοβιανούς φίλους γνωρίζοντας ότι ο δρόμος μπροστά μας είναι δύσκολος γνωρίζοντας όμως ότι είναι δυνατόν να προχωρήσουμε και να βρούμε μια λύση και το 2016 να είναι επιτέλους η χρονιά όπου η σύγκρουση αυτή θα τερματιστεί. Ευχαριστούμε πολύ την ε, κυρία Αντιπρόεδρο, η οποία βεβαίως θα παραμείνει κοντά μας και για την επόμενη συζήτηση. Να σας πω ότι έχουμε πάρει 7 προτάσεις ε, ψηφίσματος. Ε, Τώρα η συζήτηση